Dear colleagues, Dear colleagues, may we begin? Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Να σας ανακοινώσω καταρχάς ε, τις αποφάσεις των συντονιστών. Η έκθεση ίδιας πρωτοβουλία για τους whistleblowers πηγαίνει στους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ο εισηγητής θα είναι η κυρία Ροζιέρ. Αυτά περί των αποφάσεων των συντονιστών. Συνεχίζουμε τώρα με το σημείο 13. Εξέταση των τροπολογιών για την απόσπαση των εργαζομένων και ο λόγος στον κύριο Καβαντά, ο οποίος είναι και ο εισηγητής μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους ε, που συνεισέφεραν στη γνωμοδότηση αυτή στην Επιτροπή μας με τροπολογίες. Ε, σε συνέχεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων διαπιστώνω το εξής. Υπάρχουν αρκετές πολιτικές ομάδες οι οποίες ε, έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτές οι διεστάμενες απόψεις μπορούν ε, να τύχουν προσέγγισης. Ε, χωρίς να επισέλθω σε λεπτομέρειες, να σας πω ότι δεν θα συζητήσω κάποια ουσιαστικά σημεία της τροπολογίας που στόχο έχουν να αλλάξουν τη νομική βάση αυτής της πρότασης, διότι η Επιτροπή Απασχόλησης ζήτησε από την Επιτροπή μας να αποφανθεί περί της αλλαγής της νομικής βάσης η νομοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, πιστεύω ότι θα μπορούσε να είναι έτοιμη για την επόμενη συνεδρίαση ή δυνατόν για την επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει 3 και 4 Μαΐου και προτείνω να δούμε τότε αυτές τις τροπολογίες ε, για την ε, διαδικασία αυτή μετά από την προφορική παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας. Όσον αφορά τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και τις οποίες θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα, θα ήθελα να κάνω κάποιες σύντομες ε, παρατηρήσεις. Καταρχάς, ο, ο χρόνος της απόσπασης. Κάποιοι συνάδελφοι προτείνουν να διαγράψουμε ε, το χρονικό περιορισμό της απόσπασης. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι θα ήταν λογικό να περιοριστεί η διάρκεια της απόσπασης στους 6 ή 12 μήνες. Αφετέρου, η έννοια της ε, αποζημίωσης ε, λίγο πολύ η ίδια κατάσταση. Κάποιοι συνάδελφοι αναφέρονται σε αποζημίωση, κάποιοι άλλοι σε ποσοστό κατώτατου μισθού και κάποιοι άλλοι τα premium και τα επιδόματα που προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία, επίδομα μετάθεσης κλπ. Ε, επίσης αποκλείεται το ενδεχόμενο να δοθούν στα κράτη-μέλη δυνατότητες ε, να υπάρχουν κάποιες διατάξεις οι οποίες ε, θα επιοχρεώνουν τις επιχειρήσεις ε, να δίνουν συμβάσεις υπεργολαβίας οι οποίες θα υπόκειται σε συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας. Εγώ είμαι μάλλον υπέρ του θέματος γιατί είναι προφανές ότι επί των δύο αυτών θεμάτων θα μπορούσε να γίνει διαπραγμάτευση και να έχουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και με επικοδομητικό τρόπο μάλιστα. Για τις οδικές μεταφορές που είναι το τρίτο θέμα, εδώ είμαι υπέρ του να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε συγκεκριμένη νομοθεσία. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να είμαστε μάλλον επιφυλακτικοί και να μην ε, αφήσουμε το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας σε νομοθετικό κενό. Και επομένως εγώ προσωρινά μέχρι να υπάρξει συγκεκριμένο κείμενο επί του θέματος είμαι υπέρ ε, του να συμπεριληφθούν και σε αυτή την έκθεση για να μην υπάρχει κενό. Ε, επίσης για να ολοκληρώσω να πω ότι είμαι απόλυτα διατεθειμένος ε, να έχουμε αυτή την έννοια της υπόθεσης ε, εγκατάστασης εταιρείας που ε, βρίσκεται στη χώρα υποδοχής ε, του εργαζομένου ώστε να υπάρχει προστασία και αντίστοιχοι κανόνες για όλους. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα σημεία στα οποία θα ήθελα να σχολιάσω για να γνωρίζουν οι συνάδελφοι τι ακριβώς έχουμε κάνει. Thank you very much. ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καταθέσει 14 τροπολογίες και θα ήθελα να τις περιγράψω επιγραμματικά. Ο στόχος μας είναι να έχουμε έναν κανονισμό ο οποίος καλύτερα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες ε, των εργοδοτών και των απεσπασμένων εργαζομένων σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η πρόταση τελικά θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Δεν πρόκειται για τις κατασκευές, είτε τις μεταφορές, είτε οποιονδήποτε άλλον. Θαλάσσιες μεταφορές. Δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να αποκλείεται, να αποκλείονται. Πιστεύουμε ότι όλες οι μεταφορές θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. και να καλύπτεται η αποζημίωση των εργαζομένων. Στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή υπάρχει το θέμα της δημιουργίας μιας ιδιαίτερης εξέτασης για τον τομέα αυτόν. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό της αποζημίωσης. Remuneration. Αυτό δημιουργεί προβλήματα γιατί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αυτή τη στιγμή να ουσιαστικά μέσω της πρότασής της, ουσιαστικά θα αναγκάσει μάλλον τους εργοδότες να, ε, ε, να, να, να ε, ερμηνεύουν εκείνοι το εθνικό δίκαιο και αυτό πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό. Αντιθέτως, εμείς θα πρέπει να έχουμε έναν ορισμό ο οποίος να είναι ξεκάθαρος και να είναι ξεκάθαρο για τα κράτη-μέλη και με τη σειρά του τα κράτη-μέλη να ξεκαθαρίσουν στου εργοδότε μέσω τη νομοθεσία ποια είναι τα μέρη τη ε, υποζημία, τα οποία ε, ε, καλύπτονται και ποια όχι. θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ως πιθανός τρόπος υπολογισμού και ο ελάχιστος μισθός και η γεωγραφική κάλυψη και η κάλυψη κλάδων της οικονομίας. Θα πρέπει αυτά τα στοιχεία να είναι επίσης διαθέσιμα, εύκολα προσβάσιμα για να υπάρχει ισότιμος ανταγωνισμός επίσης θα προτείναμε να διαγραφεί αυτή η δυνατότητα πώς για 24 μήνες. Αυτό το όριο των 24 μηνών. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε γιατί χρειάζεται και δεν έχει προβλεφθεί κάποιο επιχείρημα ούτε από νομικής απόψεως ούτε από απόψεως ε, του γιατί να το χρειάζονται αυτό οι εργοδότες, οι αγορές, η αγορά. Υπάρχουν υπηρεσίε ε, στις οποίες ο εργαζόμενος χρειάζεται να αποσπαστεί για περισσότερους από 24 μήνες, για παράδειγμα στον τομέα των κατασκευών. Ε, τι θα κάνουμε, θα αναγκάσουμε τις επιχειρήσεις να αντικαθεστούν τους αποσπασμένους εργαζόμενους κάθε 24 μήνες. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Ε, μεταξύ άλλων, στη σχέση αυτής της οδηγίας με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό δίκαιο, στο τομέα του εργασιακού δικαίου. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει ένας σαφέστερος ορισμός της υπεργολαβίας και του αριθμό των ημερών ε, αναμήνα που αυτή τη στιγμή έχει καθοριστεί στις τρεις. Αυτές ήταν, αυτά ήταν τα κύρια στοιχεία των τροπολογιών που έχουμε προτείνει. Ελπίζω ότι ο εισηγητής θα τα λάβει υπόψη του. Σας ευχαριστούμε. Κύριο Σάγερ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι οι, τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, ως Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, διαβάζοντας τις τροπολογίες, ε, διαπιστώνω ότι έχουν υποβληθεί τροπολογίες στην Επιτροπή Γιούρη που δεν αφορούν στο, στη νομική βάση, στα νομικά ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι εναντίον ε, των προτάσεων αυτών, αλλά οι αρμοδιότητες μας ε, αφορούν τη νομική βάση. Ορισμένες σχετίζονται φυσικά και με αυτές τις τροπολογίες δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και η συνήθεια η ίδια τροπολογία να υποβάλλεται σε πολλές επιτροπές ταυτόχρονα, το έχουμε συνηθίσει αλλά όπως είπατε εμείς πρέπει να σταθούμε στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Γιούρη που είναι η νομική βάση και τα νομικά θέματα. Το σημαντικότερο νομικό ζήτημα που έχει τεθεί και έχει συζητηθεί μέχρι τώρα διεξοδικά είναι το κατά πόσον αυτή η νέα προτινόμενη οδηγία συγκρούεται με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Και εδώ πολλοί, ε, υπάρχει διχογνωμία. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν, δεν, δεν είναι συμβατές. Παλαιότερα είχα πει στην Επιτροπή ότι υπάρχει μια διάκριση, μια διαχωρισμό ανάμεσα των χωρών που είναι στη, στη, Δύση και των Ανατολικών χωρών. Από τι ε, τροπολογίε διαπιστώνω ότι αυτό δεν ισχύει. Πια ε, υπάρχουν ανησυχίε που αφορούν με, με τι διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών στον, τομέα, στον τρόπο με τον οποίο ε, οργανώνεται η συμφωνία μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων, την προστασία που υπάρχει, το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. Επομένως θα έλεγα ότι πλέον έχουμε ξεπεράσει τη σύγκρουση μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά ε, πλέον έχουμε μια πολύ περισσότερη ποικιλομορφία, ποικιλία σε σχέση με πριν, ότι, και το οποίο φαίνεται από τις τροπολογίες. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ορισμένα κράτη-μέλη που είναι εκείνα τα οποία προστατεύουν τους εργαζόμενούς τους πιο αποτελεσματικά από όμορες χώρες, από γειτονικέ τους χώρες, είναι εκείνα τα οποία έχουν, ε, τους δημιουργείται πρόβλημα με αυτή την πρόταση της Επιτροπής. Ένα άλλο θέμα το οποίο κατά την άποψή μου παραμένει ε, προβληματικό είναι αυτός ο κανόνας των 24 μηνών το, ο οποίος δημιουργεί προβλήματα και σε σχέση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, γιατί δημιουργείται ε, μια νέα έννοια στο δίκαιο, το οποίο, η οποία δεν υπήρχε μέχρι στιγμή και η οποία σου δημιουργήσει νέες ε, δυσκολίες, προσπαθώντας να αποφύγει άλλες. Και πιστεύω ότι αυτή η πρόβλεψη αντίκειται ακριβώς στην ελευθερία ε, παροχής υπηρεσιών. Υπευλήθησαν τροπολογίες προσπαθώντας να το διορθώσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι επί τους ουσίες στη ρίζα της αυτή η πρόταση για τους 24 μήνες ε, δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα όσον αφορά τους ορισμούς, έχουμε τον ορισμό της αποζημίωσης και το πώς αυτό ε, συνδυάζεται με την έννοια του μισθού. Ε, Έχουμε μια σειρά προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εάν αυτοί οι δύο ορισμοί συμπίπτουν και μια άλλη σειρά προβλημάτων που θα παρουσιαστούν εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ αυτών των δύο ορισμών. Εάν συμπίπτουν αυτές οι δύο έννοιες δεν υπάρχει κανένας λόγος να δημιουργήσουμε νέες, ε, νέα ορολογία που να δημιουργεί σύνθεση, σύγχυση. Εάν πάλι υπάρχουν διαφορές, οι διαφορές αυτές δεν είναι καθόλου ξεκάθαρες από αυτή την προτινόμενη οδηγία. και πρόκειται ήδη για έναν τομέα του εργατικού δικαίου που είναι προβληματικός, δηλαδή που έχει ε, αμφισημίες. Θα υποστηρίξω λοιπόν τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μεγάλη ε, ανησυχία και τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Ε, και έχουμε υποβάλει ε, τροπολογίες σχετικές. Έχουμε ζητήσει και γνωμοδότηση της Νομικής Επιτροπής. Ε, και δυστυχώς το, ακριβώς το ζήτημα ε, το οποίο μας απασχολεί και για το οποίο ζητήσαμε τη γνωμοδότηση ήταν εκείνο που παρέμεινε ασαφές στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Ε, εμείς πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε το αίτημα, την έννοια του αιτήματος απασχόλησης, Θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν την πρόταση που μας έχει έρθει από την Επιτροπή ε... Απασχόλησης και από τη δικιά μας πλευρά, από την πλευρά της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, καλό θα είναι η νομική μας ε, γνωμοδότηση, η, η, η θέση που θα λάβουμε από νομική απόψεως να είναι ξεκάθαρη, έτσι ώστε μετά η συζήτηση στην Επιτροπή Αποσχόλησης ή και στην Ολομέλεια να μπορεί να προχωρήσει όπως πρέπει. Σας ευχαριστούμε κυρία Τελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Καβαντά, και να τον ενθαρρύνω να συνεχίσει να είναι αισιόδοξο. Συμφωνώ ότι ε, θα πρέπει να καθυστερήσουμε τη συζήτηση για τη νομική βάση, να την κάνουμε σε άλλη συνεδρίαση, γιατί περιμένουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, η οποία έχει ζητηθεί ούτως ή άλλως επισήμως. Ε, πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να δούμε και τι θα περιμένουμε και άλλες επιτροπές για το θέμα αυτό, αλλά ε, οι τροπολογίες μου θέλουν να δώσουν στην οδηγία δύο βάσεις. Δηλαδή, και νομίζω ότι πέραν των τεχνικών ε, και νομικών θεμάτων είναι και πολιτικό. Le η πρόκληση είναι να αποδείξουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών δεν αντιβαίνουν στο ε, εργασιακό δίκαιο και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Διότι πολλές φορές μας λένε ότι ασχολούμαστε μόνο με την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και υπηρεσιών και ότι δεν ε, λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες ε, και την ευημερία των ανθρώπων. Για μένα ε, ακριβώς ε, αυτό ε, επιθυμούμε να κάνουμε. Στο ίδιο κράτος μέλος οι εργαζόμενοι που κάνουν την ίδια δουλειά να την χάνουν ίσης μεταχείρισης. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλη πρόκληση και πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά τι θα πούμε και τι θα δηλώσουμε σε σχέση με την κοινή γνώμη. Δεν θέλουμε να... Ε, θέσουμε σε δύσκολη θέση ένα πάροχο υπηρεσιών. Ίσα ίσα θέλουμε ε, να έχει ίσους όρους εργασίας ένας εργαζόμενος που ζει σε μια χώρα και κάποιος ο οποίος αποσπάται σε αυτή τη χώρα για να εργαστεί. Ε, θα περιμένω βεβαίως τη συζήτηση η οποία θα γίνει σίγουρα την επόμενη φορά αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποδείξουμε ότι υπάρχουν δύο νομικές βάσεις. Δεν μπορούμε να ε, δώσουμε βαρύτητα μόνο σε μία. Κατά τα άλλα, για τις υπόλοιπες τροπολογίες, νομίζω ότι το κριτήριο της αποζημίωσης είναι σημαντικό. Εμείς εδώ σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στους κανόνες ενός κράτους μέλους που καθορίζει τα θέματα των μισθών και επομένως ε, θεωρούμε ότι αυτή είναι ε, αρμοδιότητα του κράτους μέλους αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν ε, τη μισθολογική αποζημίωση ε, και ό,τι υπαγορεύει ο νόμος, αλλά και ό,τι προκύπτει από τις λογικές διαπραγματεύσεις. Ε, όσον αφορά τη διάρκεια, εδώ είμαι αρκετά αισιόδοξη. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη διάρκεια. Αλλά να πω ότι 24 μήνες μου φαίνεται μεγάλο διάστημα. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε προτείνει ε, μικρότερο διάστημα απόσπασης. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι ε, αυτά είναι τα ουσιαστικά από τι ε, τροπολογίες και αν ε, συμφωνήσω και εγώ με την αισιοδοξία του κυρίου Καβαντά, σίγουρα θα βρούμε μια λύση, ένα συμβιβασμό, χωρί να χάσουμε ε, και τις βασικές αρχές που υπερασπιζόμαστε. Δηλαδή, την νομιμότητα και το σεβασμό προ τον οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγή του και τη δουλειά του η οποία επηρεάζεται από αυτούς τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ο κύριος Άντερσον. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω κι εγώ ευχαριστώντας τον εισηγητή. Δεν θα συζητήσουμε σήμερα τη νομική βάση. Αλλά έχω και καταθέσει σχετική τροπολογία. Θα περιμένουμε για αυτή τη συζήτηση. Η ουσία αυτής της οδηγίας είναι να έχουμε καλύτερη αγορά εργασίας. Θέλουμε να δώσουμε στους εργαζομένους και στις επιχειρήσεις ευκαιρίες και να αυξήσουμε τις ελευθερίες τους. Δεν ε, θα πρέπει να είναι ένας τρόπος για να αποφύγουμε την ομοθεσία και να εκμεταλλευόμαστε τους εργαζομένους. Αυτή είναι η ουσία αυτής της οδηγίας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία λύση που όντως ε, θα επιδιεχάνει αυτό. Όσον αφορά τα θέματα της ε, αυθεντικής απόσπασης, ε, ε, ελπίζουμε ότι οι αποσπάσεις είναι όντως αυθεντικές και έχουμε και καταθέσει σχετικές τροπολογίες και αυτό σημαίνει ότι αν διαπιστώνεται ότι κάποιος δεν είναι πραγματικά αποσπασμένος, τότε θα πρέπει να ισχύει η νομοθεσία της χώρε θα πρέπει να είναι προβλέψιμο το αποτέλεσμα δηλαδή ε, και αυτό είναι λογικό εκτός ε, δεδομένου ότι μπορεί να ευνοείται από την νομοθεσία αν θεωρείται αποσπασμένος. Αυτό είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι τα συστήματα της αγοράς εργασίας των κρατών μελών είναι πάρα πολύ διαφορετικά και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Σε κάποιες χώρες υπάρχει πρόγραμμα κατώτατου μισθού, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Και η οδηγία αυτή πρέπει να ε, λειτουργεί ανεξάρτητα από το σύστημα που διαθέτει το κάθε κράτος μέλος και ε, έχω κάποιες τροπολογίες οι οποίες θα λύσουν αυτό το πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη. Τροπολογία που λέει ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίσουν κανόνες για τις μυθολογικές αποζημιώσεις βάση του δικαίου τους. Ε, μπορεί να σας φαίνεται ίσονο σημασία στη λεπτομέρεια, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική για τις χώρες που έχουν συλλογικές συμβάσεις. Όσον αφορά το χρονικό όριο, εγώ θεωρώ ότι έξι μήνες είναι λίγοι. Γι' αυτό και υπέβαλα τροπολογία για 12 μήνες. Μια συμβαστική λύση. και προσβλέπω στην συνέχεια της συζήτησης για το θέμα αυτό. much. Mr. Foss. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να θίξω δύο σημεία εν συντομία που έχουν να κάνουν με την νομική περιπλοκή του ζητήματος. θα πρέπει να αναλάβουμε υπόψη μας ε, ότι δεν μπορούμε να επέμβουμε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις των κρατών μελών. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικά, διαφορετικές συνταγματικές προσεγγίσεις και δεν πρέπει με αυτόν τον τρόπο να μπούμε στα πόδια των κρατών μελών. Μετά από αυτούς τους 24 μήνες, να πω επίσης, ε, για τους 24 μήνες να πω ότι θα πρέπει να προσέχουμε ε, ότι θα πρέπει να, να υπάρχει ελευθερία για κάποια σύμβαση, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για να μην φτάσουμε σε μια περίεργη κατάσταση ε, όπου ένα κράτος μέλος, ένα κράτος δικαίου θα υπόκειται σε δυσκολίες και θα πρέπει κάποιος να υπόκειται στην πατρίδα του, ας πούμε ποια είναι η Αυστρία και τελικά να έχει αποσπαστεί στη Γερμανία και ένα αυστριακό δικαστήριο να πρέπει να δικάσει την απόφαση, μια υπόθεση που σχετίζεται με τη δική του σύμβαση. Μετά από 24 μήνες λοιπόν είναι πολύ δύσκολο θεωρώ να, ε, να λύσουμε το ζήτημα, ειδικά μπορεί να φτάσουμε σε περίεργες καταστάσεις αν το ένα κράτος πρέπει να προσφύγει ε, κατά ενός άλλου κτλ. Πρέπει να τα σκεφτούμε αυτά. Thank you, Mrs. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό μου η συζήτηση ε, για την οδηγία για τις αποσπάσεις μου θυμίζει και τη συζήτηση με το κοινωνικό dumping. Είχαμε μια επιτροπή ακρόσεις στο Παναμα, για τον Παναμά η οποία είχε ακριβώς ασχοληθεί με την φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή γενικά ε, φαίνεται ότι κάποιοι έδιναν μισθούς ε, που οδηγούσαν σε κοινωνικό ντάμπινγκ για να αποφύγουν φορολογία. Ε, το ίδιο ισχύει και εδώ με τις εικονικές εταιρείες που υπάρχουν για να μην μπορούν να μην πληρώνουν τις σωστές αποζημιώσεις, τη σωστό μισθό. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ίση αμοιβή για ίση εργασία. Έχει να κάνει ε, λοιπόν το θέμα αυτό όχι μόνο με τη διαμόρφωση των μισθών αλλά και με τα δικαιώματα τα εργασιακά. Θα πρέπει να έχουμε κάποια ελάχιστα στάνταρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλουμε όλοι να προχωρήσει αυτό να γίνουν πιο μικρές οι διαφορές ε, μεταξύ των κρατών. Όμως αυτό δεν ισχύει ακόμα και γι' αυτό οι τροπολογίες μας ε, προσπαθούν στην ουσία να οδηγήσουν ε, στο να αποφύγουμε αυτό το forum shopping, να προσπαθεί κανείς να βρει το σύστημα στο οποίο θα πρέπει να τηρεί τα λιγότερα στάνταρ για την ελευθερία παροχής υπηρεσιών τώρα. Φυσικά είναι μία από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες που πρέπει να σεβόμαστε, όμως υπάρχει και μεγάλη ε, κατάχρησή της. Σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου πολλές φορές ε, δεν έχει να κάνει με την παροχή μιας υπηρεσίας, αλλά πολύ συχνά με την ε, παράκαμψη ότι σε επίπεδο ουσιαστικού ε, δικαίου θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορισμός ενός, ε, ε, του, της λέξης απασχολούμενος. Υπάλληλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε λοιπόν και αυτό το στοιχείο σε επίπεδο νομικό. Και γι' αυτό υπάρχουν οι τροπολογίες ε, που ε, θέλουν ακριβώς να τραβήξουν μια ξεκάθαρη γραμμή εκεί. Ότι πρέπει να μπορεί να παρέχεται ελεύθερα μια υπηρεσία, αλλά να μην χρησιμοποιείται αυτό ως παράκαμψη της νομοθεσίας. Να πω επίσης ε, κάποια πράγματα για τους δανειζόμενους υπαλλήλους όπως τους αναφέρουμε στα γερμανικά, Leiharbeiter, είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωστή ε, αντιμετώπιση. Έχουμε κάποια τέτοια ε, νομοθεσία ε, για τους εργάτες υποδανισμό που μπορούν να πηγαίνουν από τη μία χώρα στην άλλη έτσι ώστε να έχουν την ίση μεταχείριση και να είναι ξεκάθαρο ε, αυτό ε, το σημείο, κατέθεσα τις αντίστοιχες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και εγώ δύο παρατηρήσεις. Η μία που έχει να κάνει με το κοινωνικό dumping Μέσα στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας ε, η έννοια της ίσης αμοιβή για ίση εργασία είναι εντάξει, όμως θεωρώ ότι στο ευρύτερο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των εργαζομένων θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε και την αρχή της ίσης αμοιβή για ίση εργασία σε ίση επιχείρηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί βλέπουμε διακρατικές εταιρείε να οργανώνουν κοινωνικό dumping. Η ίδια δουλειά αμοιβεται διαφορετικά στο κάθε κράτος μέλος. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή ιδέα. Έχουμε την πολύ γνωστή υπόθεση της Σαμπένα από το παρελθόν. Τώρα αν θα, εξαιρεθεί, θα εξαιρεθούν οι μεταφορές από το πλαίσιο της οδηγίας, εγώ θεωρώ ότι αν εξαιρεθούν δεν είναι μόνο κίνητρο για την ε, Επιτροπή να κάνει ένα πιο συγκεκριμένο νομοθετικό σχέδιο, αλλά θα ηρεμήσει λίγο και τις ανησυχίες των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Ο κύριος Λεμπρετών τώρα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ ξεκάθαρος. Από την πλευρά του Front National είναι καταδικάσιμη αυτή η οδηγία γιατί είναι κοινωνικό ντάμπινγκ εντός της ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει παραγάγει καταστροφικές επιπτώσεις στην χώρα μου όπου έχουμε 6.000 ε, αποσπασμένους ε, σε θέσεις που θα μπορούσαν να καταλαμβάνουν Γάλλοι. Η κοινή γνώμη στη Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι διχασμένη και γι' αυτό ε, δυστυχώς είναι επίγον το θέμα σήμερα. Δεν θέλω σήμερα να καταθέσω καμία τροπολογία γιατί δεν θέλω να συνεισφέρω σε αυτή την προσπάθεια τελευταία στιγμή να σωθούν όσα μπορούμε. Έχω δύο βασικές και ουσιαστικές ε, παρατηρήσεις. Μία για την ισότητα της αμοιβή. Σήμερα στην πρόταση αναφερθήκατε σε αυτό. Ε, το ελάχιστο είναι ε, να έχει ένας αποσπασμένος εργαζόμενος την ίδια αμοιβή με έναν μη αποσπασμένο αυτό θα βοηθούσε σε κάποιο βαθμό να αποφύγουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ. Όμως πρέπει να σεβόμαστε γενικά τις συνθήκες για την αμοιβή, αμοιβή των εργαζομένων. Για την διάρκεια τώρα θεωρώ ότι ε, είναι καλή ιδέα Έξι μήνες με δύο χρόνια προτείνεται. Όσο λιγότερο για μένα θα ήταν το βελτιστό, γιατί έτσι θα δείξουμε ε, το προσωρινό χαρακτήρα αυτής ε, της εργασίας ε, και νομίζω ότι συνάδει με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, γιατί η Ευρώπη δεν είναι σε καμία περίπτωση μια κοινωνική Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε λίγο να βελτιώσουμε αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε καν αυτοί οι αποσπασμένοι πάλι να υπάρχουν κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Σάιερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη που δεν ευχαρίστησα τον εισηγητή στην αρχή. Ήμουν λίγο αγενής, αλλά έτρεχα μεταξύ διαφόρων επιτροπών. Το διορθώνω τώρα. Ζητώ το λόγο, όχι γι' αυτό βέβαια, δεν είναι θέμα πρωτοκόλλου, αλλά θέλω να πω στην κυρία Ρέγνερ ότι αυτή η συζήτηση και σε μένα θυμίζει τη συζήτηση για το κοινωνικό dumping. Το θέμα της παράκαμψης και της κατάχρησης είναι πράγματα που με ε, αφορούν και μαγγίζουν. Ε, οι νέοι κανονισμοί συνήθως προσπαθούν να διορθώσουν κάτι, ε, να το να απογορέψεις την όλη διαδικασία για να αποφύγεις αυτή την κατάχρηση και την παράκαμψη δεν είναι σωστό. Κατά τη γνώμη μου, ο περιορισμός των δύο ετών, γιατί ως τώρα δεν έχουμε περιορισμό, είναι στην ουσία ένας τρόπος να σταματήσουμε μετά από δύο χρόνια την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ίσως είναι λίγο κατηγορηματικός ο τρόπος που το θέτω, αλλά αυτό είναι. Ως τώρα δεν το είχαμε, από εδώ και πέρα θα το έχουμε και είναι περιορισμός. Είναι, ας πούμε, σαν ε, να έχουμε κάποιους που δεν αγοράζουν εισιτήριο στο τρένο όταν ανεβαίνουν για να το χρησιμοποιήσουν και επειδή το κάνουν αυτοί εμείς ε, στην ουσία τιμωρούμε όλους τους επιβάτες. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Πάντοτε υπάρχουν καταχρήσεις των κανόνων και για να το αποφύγουμε υπάρχουν πιο εξελιγμένοι τρόποι. Μπορεί να έχουμε ας πούμε καλύτερο έλεγχο των κανονισμών όχι να σκοτώνουμε την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Ξέρουμε το κοινωνικό υπόβαθρο αυτής της κατάστασης. Έχω ε, δυσκολία να καταλάβω ε, λέξεις όπως ε, μάχη που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι. Είναι σαν να λέμε για την πυρηνική βόμβα κατά του Άισις. Ε, κάτι τέτοιο κάνουμε και εδώ. Χρησιμοποιούμε μια πυρηνική βόμβα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων θα πρέπει να εξετάσουμε καλύτερα την συνθήκη, την νομική βάση και την αρχή της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε. Και για να μην αφήσουμε απ' έξω το κοινωνικό κομμάτι, να πω ότι Υπάρχουν ε, δυνάμεις στην Ευρώπη που θέλουν να σταματήσουν κάθε είδους ελεύθερη διακίνηση εργασίας. Τα έχουμε ακούσει αυτά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να γίνουμε αρρωγοί σε τέτοιες καταστάσεις. Η κυρία Ροζιέρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την ξεκάθαρη παρουσίαση των διακευευμάτων αυτού του κειμένου γιατί είχαμε λίγο φύγει ε, στην αρχή της συζήτησης από το θέμα, αλλά τώρα με τα σχόλια των ε, συναδέλφων έχουμε φύγει ακόμα παραπέρα από την καρδιά της συζήτησης. Αυτή η οδηγία δεν προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, επιτρέπει ας πούμε σε κάποιους εργαζομένους που ζουν σε μια χώρα διαφορετική από τη χώρα προέλευσής τους να ε, χρησιμοποιήσουν για μικρό χρονικό διάστημα τα δικαιώματα που είχαν στη χώρα προέλευσης. Αυτό στην ουσία είναι για να εγγυηθεί δικαιώματα στους ε, μισθωτούς. Αυτό όμως ε, δυστυχώς που συμβαίνει είναι ότι χρησιμοποιείται διαφορετικά από τον αρχικό της στόχο που ήταν η προστασία για να οργανωθεί μια, ένας κοινωνικός ανταγωνισμός και κάποιοι μισθωτοί που έχουν ε, αποσπαστεί σε κάποιες ε, χώρες στην ουσία να μην χαίρουν των δικαιωμάτων που έχουν οι ντόπιοι. Αυτό είναι το έλλειμμα της οδηγίας. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν να χρησιμοποιείται η οδηγία για να υπάρχει αυτός ο κοινωνικός ανταγωνισμός. Τώρα τα θύματα είναι οι εργαζόμενοι και στην χώρα ε, καταγωγής και στη χώρα ε, προορισμού. Γιατί κανείς δεν χαίρεται των δικαιωμάτων που δικαιούται. Στην ουσία η οδηγία χρησιμοποιείται για να στερηθούν οι άνθρωποι αυτοί τα δικαιώματά τους. Είχα την δυνατότητα να συζητήσω με μαθητευόμενους ε, στις κατασκευές που είναι ένας από τους βασικούς τομείς που πλήττεται και λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί τους στέρουν ένα κομμάτι της δουλειάς τους, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι ίδιοι θύματα αυτών των παρακάψεων. Είναι λοιπόν εδώ η ώρα να αποφύγουμε μια κακή ε, χρήση μιας οδηγίας και να αποφύγουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των εργαζομένων, με το χάσμα μεταξύ μισθών και με την κακή χρήση ε, μιας ε, νομοθεσίας για να μειωθεί ο μισθός των ανθρώπων στην ουσία. Μιλάμε για το ανταγωνισμό. Αυτά που αναφερθήκανε ε, έχουν να κάνουν στην ουσία και με την, την οδηγία για τις υπηρεσίες, για την ελεύθερη χρήση των υπηρεσιών, που έχει να κάνει ε, με εταιρείε οι οποίε ε, στην ουσία συγχαίουν δύο ιδιότητε, είναι και εταιρείε, είναι και μισθωτοί και εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά που ε, υπόθηκαν στην αρχή τη συζήτηση είναι αυτά που έχουν πραγματικά να κάνουν τη συζήτηση και θα μα οδηγήσουν στο σωστό αποτέλεσμα για να αποφύγουμε αυτό που είδαμε στην καρικατούρα της Ευρωπαϊκή Ένωσης που παρουσιάζεται σαν να κοιτάζει μόνο το θέμα τη ελεύθερη αγορά και όχι τα δικαιώματα των ε, εργαζομένων. Η κυρία Ρέγνερ, ευχαριστώ. Ε, θα ήθελα και εγώ ε, να συμπληρώσω λίγο αυτό που μόλις είπε η κυρία Ροζιέρ. χαίρομαι πολύ που ο κύριος Καβαντά αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις οδικές μεταφορές γιατί υπάρχουν φυσικά πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα προβλήματα να πω ένα παράδειγμα στη δική μου χώρα δεν είναι ε, μία εξαίρεση εδώ, ε, ε, τα μαύρα πρόβατα που έχουμε συνήθως. Έχουμε στις οδικές ε, μεταφορές μια εταιρεία η οποία έχει την έδρα και τις ε, δραστηριότητες της ε, στην Αυστρία όμως έχει ιδρύσει και μια άλλη εταιρεία σε μια άλλη χώρα με δανεικούς εργαζομένους κάνει εκεί τις συμβάσεις ουσιαστικά λοιπόν ο υπάλληλος πληρεί την τον ορισμό του εργαζομένου ε, του υπαλλήλου. Απ' την άλλη όμως έχει και μία σύμβαση η οποία τον υποχρεώνει να χρησιμοποιεί την ελευθερία ε, παροχής υπηρεσιών όταν παρέχει υπηρεσίες στην Αυστρία και η οδηγία για την απασχόληση στην ουσία με αυτό το θέμα ασχολείται. Να μην επιτρέπεται σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου αυτό το πράγμα και όταν υπάρχουν κατάχρηση ε, μέσα από εικονικές ε, αποσπάσεις αυτό να αντιμετωπίζεται. Αυτό το θέμα το έχουμε συζητήσει ε, πολλές φορές και πρέπει να το περιορίσουμε μέσα στα πλαίσια αυτής της οδηγίας. Να μην μπερδεύουμε την ελευθερία της υπηρεσίας με την ελευθερία της απόσπασης. Κυρία Ράγκνερ, λέει ο Πρόεδρος, ε, έμεσα υποστηρίξατε αυτό που είπα πριν. Ίση αμοιβή για ίση εργασία στην ίδια επιχείρηση κυρία Ροζιέρ, να πω ότι εμέρη διαφωνώ, διότι θεωρώ αυτά, ότι αυτά τα θέματα πρέπει να τα ε, εξετάζουμε μέσα στο ε, ευρύτερο πλαίσιο των τεσσάρων ελευθεριών της αγοράς. Αυτό που συζητούμε τώρα έχει να κάνει με τη δυνατότητα εταιριών από ε, άλλες χώρες να ανταγωνιστούν σε επίπεδο μισθολογικό. Είναι κατά του δικαιώματος αυτών των εταιριών να έχουν πρόσβαση στην αγορά ενός άλλου κράτους μέλους. Εμπόριο και πρόσβαση στην αγορά. Ας δούμε λοιπόν την ευρύτερη εικόνα, είναι καλύτερος τρόπος. Η Επιτροπή θα ήθελε να πάρει το λόγο. Merci. Merci, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω γαλλικά. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ξεκινώ ευχαριστώντα και ε, συγχαίροντα τον εισηγητή σα για το προσχέδιο έκθεσης που έχει παρουσιάσει, το οποίο θεωρούμε ότι είναι σωστά ισορροπημένο και ε, έχει θέσει το δάκτυλο με τον τύπο των ήλων σε ένα σύντημα το οποίο ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο. Είναι, είναι θέματα ε, θα ήθελα να σας παρουσιάσω μάλλον κάποιες ιδέες οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν γενικά τη συζήτησή σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι η εξή. Ένα σύνολο τροπολογιών, είτε του εισηγητή είτε μελών, προσπαθούν να βελτιώσουν την, α, το κείμενο για να γίνει πιο ξεκάθαρο, το κείμενο που έχει προτείνει η Επιτροπή για να γίνει πιο ξεκάθαρο. Και αυτές τις τροπολογίες τις καλωσορίζουμε οποιαδήποτε βελτίωση ε, που συνεισφέρει στην ασφάλεια δικαίου και στη σαφήνεια του κειμένου είναι καλοδαχούμενη. Για παράδειγμα, οι προτάσεις που συμπεριλαμβάνουν τον ελάχιστο κατώτατο μισθό στην αποζημίωση. Γιατί, όπως υπόθηκε, η έννοια του του μισθού δεν είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι ξεκάθαρο δηλαδή να καθορίσουμε σε κάθε κράτος μέλος τι συνιστά κατώτατο μισθό στην πράξη. Ε, παρά το γεγονό ότι ε, κάποια κράτη-μέλη στη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έλαβαν μέτρα προστατευτικά προς τους εργαζόμενους, στην πράξη ε, διαπιστώνουμε κάτι διαφορετικό να γίνεται. και διαπιστώνουμε ότι οι τροπολογίε που έχουν προτείνει και ο συγητή σα και μέλη τη Επιτροπή σα πηγαίνουν προ αυτή την κατεύθυνση και τι ε, καλωσορίζουμε. Είμαστε θετικά απέναντί του. Σε αντίθεση με αυτό που υπόθηκε, ε, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει κανέναν περιορισμό στην απόσπαση. Χρονικό περιορισμό. Δεν προτείνουμε να περιορίζεται η απόσπαση στους 24 μήνες. Ε, ίσως αυτό να δίνεται μια εικόνα προσπαθώντας εν τη του λόγου του κάποιος να παρουσιάσει την, την ε, οδηγία, αλλά δεν ισχύει. Η ε, οδηγία προβλέπει ότι η απόσπαση μπορεί να διαρκεί για όση διάρκεια χρειάζεται για την παροχή της υπηρεσίας. 26 μήνες ή όσους χρειάζεται. Δεν υπάρχει κάποιο όριο. Αυτό που λέμε αντιθέτως είναι ότι όταν αυτή η απόσπαση προβλέπε, να ξεπεράσει τους 24 μήνες είτε επί της ουσίας, επί, της πράγματι ξεπερνά τους 24 μήνες, τότε το κράτος μέλος ε, προορισμού του αποσπασμένου εργαζόμενου γίνεται, καθίσταται το κράτος στο οποίο ε, έχει την ε, εργασία του ο εργαζόμενο και άρα εφαρμόζεται το εργατικό δίκαιο του, του κράτου μέλου προορισμού. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τη απόσπαση που ξεπερνά τις 24 μήνε και τη απόσπαση που είναι ε, πιο σύντομη τι είναι η πρόβληση, πρόβλεψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προσπάθησε να θέσει κάποιο όριο στο χρονικό στην απόσπαση. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με το πνεύμα της οδηγίας και επίσης με τη συνθήκη. Απλώς προσπαθούμε να θέσουμε κάποιους ε, όρους για τις περιπτώσεις εκείνες που η απόσπαση ξεπερνάει τους 24 μήνες. Ε, δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, κάποιες ακόμα μικρές παρατηρήσεις έχω να κάνω. Όσον αφορά τη διαφάνεια, ε, που ανέφεραν, ένα θέμα που ανέφεραν ορισμένοι βουλευτέ. Ε, είναι προφανές ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ε, έχουν ανάγκη να, υπάρχει πλήρης διαφάνεια γιατί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε, ένα νέο κράτος μέλος που δεν γνωρίζουν και αντιστοίχω και οι εργαζόμενοι χρειάζεται να γνωρίζουν όλα τα ε, στοιχεία που αφορούν στον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν Ποιε είναι οι αρμόδιε αρχέ για την επιθεώρηση εργασία, για παράδειγμα, οι όροι κτλ. Ε, ε, γνωρίζετε ότι ήδη στο άρθρο 5 της οδηγίας του 2014 τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν τους αποσπασμένους εργαζόμενους ε, για το εργατικό δικαίωμα και ιδιαίτερα για τις συλλογικέ συμβάσεις. Είναι στο άρθρο 5 της οδηγίας του 2014 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλωσορίσει οποιαδήποτε πρόταση τροπολογία, τροποποίηση ε, η οποία θα αυξήσει τη διαφάνεια και τα στοιχεία που δίνονται για τους όρους εργασίας ε, που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος. Αυτό φυσικά δημιουργεί αυξημένο διαχειριστικό φόρτο ε, για τα κράτη-μέλη ε, που αποδέχονται ε, προορισμού, που αποδέχονται υπεσπασμένους εργαζόμενους, αλλά αξίζει αυτή η επιπλέον προσπάθεια γιατί θα έχουν περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι. Και τέλος, η οδηγία του 2014 και ο στόχος της πρότασης της Επιτροπής δεν είναι, μάλλον η πρώτη μας, η, η, τωρινή δεν είναι να βελτιωθεί ο τρόπος εφαρμογής των κανόνων. Αυτό καλύπτεται από την οδηγία του 14. Δεν οπισθοχωρούμε καθόλου. Και το επισημαίνω αυτό, γιατί ορισμένες τροπολογίες πηγαίνουν προς εκείνη την κατεύθυνση και αυτό μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι οι προβλέψεις της οδηγίας του 2014 δεν ήταν επαρκείς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε στοιχεία που να το δω. αποδεικνύουν αυτό. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι ακριβώ αυτό που αναφέρεται στο κείμενο, είναι η όρια εργασία των αποσπασμένων εργαζομένων και σε αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε και να περιοριστούμε. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη μια ερώτηση προς τον εισηγητή για το χρονοδιάγραμμα. Εδώ στις σημειώσεις μου βλέπω ότι η έγκριση στην Επιτροπή προβλέπεται για 30 Μαΐου. Αλλά υπάρχει δυνατότητα να αναβληθεί και για τις 20 Ιουνίου. Ο κύριος Καβαντά εξακολουθεί να μένει στις 30 Μαΐου. Υπολογίζεται ότι θα το τελειώσετε εκεί. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σήμερα. Τέλος εβδομάδας, αν δεν σας πειράζει. Και μιας και έχω και το λόγο, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ επαγγελματικό το κλίμα στο θέμα αυτό. Ούτως ή άλλως η πρόταση είναι και το πλέον κατάλληλο μέσο και εδράζεται σε ρεαλιστικές βάσεις. Επομένως, ε, προσβλέπω και στη συνεργασία με τους συναδέλφους για να ολοκληρώσω την ε, γνωμοδότηση αυτή και Ακόμα και όταν τα πράγματα είναι ιδεχθή, θα ήθελα να πω στον κύριο Σβόβαθα το γεγονός ότι συμφωνείτε με την κυρία Ρέγνερ με γέμισε αγάπη, χαρά και δεν είναι και η πρώτη φορά που το επισημαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, ολοκληρώθηκε το σημείο 13 και συνεχίζουμε με το σημείο 12 εξέταση των τροπολογιών για τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενέα αγορά και δίνουμε το λόγο στην κυρία Λεγκρίπ, η οποία είναι η συγγήτρια. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω, σήμερα το πρωί πρέπει να συζητήσουμε και τις τροπολογίες που υπευλήθησαν για το σχέδιο γνωμοδότησής μου για τις ε, διαδικτυακές πλατφόρμες ε, στην ψηφιακή ενή αγορά ε, μία γνωμοδότηση ε, την οποία συντάσσουμε για την Επιτροπή Ήτρε και την Επιτροπή ΕΙΜΚΟ, που είναι οι δύο αρμόδιες επί της ουσίας ε, επιτροπές. 81 τροπολογίες κατατέθηκαν το σύνολο. Πρέπει να πω ότι και εγώ ίδια τελικά διόγκωσα τον αριθμό των τροπολογιών, γιατί υπέβαλα περίπου 15 τροπολογίες διόρθωσα τον εαυτό μου με στόχο να διευκρινίσω λίγο την αρχική μου πρόταση και να συμπληρώσω, να εμπλουτίσω το κείμενο του σχεδίου της νομοδότησης που είχα υποβάλει αρχικά πριν από κάποιες εβδομάδες. Οι διάφορες τροπολογίες ε, που υπευλήθησαν από τους και ηγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους και τους οποίους ευχαριστώ ε, αφορούν ε, μια πλειάδα θεμάτων, όλα ενδιαφέροντα για σήμερα θα σταθώ σε κάποια βασικά θέματα για τα οποία υπάρχει σύγκληση σε ένα τμήμα των τροπολογιών που κατατέθησαν και είναι en ligne dans digital single market. Euh, les sujets το πώς διαρθρώνεται αυτή η γνωμοδότηση για την ψηφιακή αγορά και τις διαδικτυακές πλατφόρμες ε, και να αναφερθώ και σε ένα θέμα το οποίο ε, είχε πολλές τροπολογίες, ο ορισμός αυτής της πλατφόρμας ε, και το πώς μπορούμε να τα συμπεριλάβουμε σε ένα νομικό πλαίσιο, το θέμα του, σε ευθύνη των ε, δομών αυτών ε, και τα θέματα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, το νομικά ζητήματα κατά του συγκεκριμένου αμφισβητούμενο περιεχομένου. Είναι πολύ σημαντική και αυτή η έννοια και επίσης ε, ε, οι σχέσεις B2B μεταξύ των επιχειρήσεων για τις πλατφόρμες, ε, τη σχέση που έχει η πλατφόρμα με τον εμπορικό εταίρο του Υπήρξαν κάποιες ενδιαφέρουσε τροπολογίες για τη σημασία της ε, διαχείρισης των δεδομένων και της διαφάνειας των αλγορίθμων, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφέρω εδώ όλες τις τροπολογίες που κατατέθησαν. Όσον αφορά τον ορισμό της πλατφόρμας, ε, ε, γιατί προσφέρουν μια ποικιλία ε, υπηρεσιών, είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα αυτό και εκεί υπάρχουν αρκετές συνεισφορές. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ώστε να υπάρξει μια προσέγγιση απόψεων, να υπάρχουν αρκετές τροπολογίες ε, στις οποίες υπάρχει μια αντίστοιχη κατεύθυνση και απλώς επιθυμείται μια διευκρίνηση για το τι ακριβώς είναι αυτές οι πλατφόρμες. Και επίση για ένα θέμα το οποίο μας φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον, όσον αφορά την ευθύνη ε, για τις πλατφόρμες, είχαμε αρκετές τροπολογίες και μεγάλη σύγκληση απόψεων, επομένως αρκετά μεγάλη πλειοψηφία ε, στις τροπολογίες που υπευλήθησαν για το θέμα αυτό που προσπαθούν και αυτές να διευκρινίσουν την ευθύνη που έχουν αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες σε πολλά θέματα και χαίρομαι που υπάρχει σύγκληση απόψεων της πλειοψηφίας ε, για να μπορέσουμε να ορίσουμε και τις πλατφόρμες αλλά και την ευθύνη που φέρουν και θα στηριχτώ σε αυτή τη σύγκληση απόψεων και χαίρομαι που αρκετοί συνάδελφοι συμφωνούν με την ιδέα να υπάρχει η έννοια της διαφάνειας και της ισοτιμίας στις διάφορες πρακτικές και στις ε, δραστηριότητες ε, που έχουν αυτές οι διαδικτυακές πλατφόρμες. Δεν θα μακρηγορήσω. Όσον αφορά το θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και της διανοητικής ιδιοκτησίας, εδώ έχουμε αρκετές τροπολογίες οι οποίες ε, πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση που θέλησα να πάω και εγώ στο σχέδιο γνωμοδότηση ε, και σε κάποιες από τις τροπολογίες μου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό φυσικά ε, απηχεί και κάποιες ε, συζητήσεις που είχαμε σε άλλα θέματα, σε άλλα νομοθετικά έργα, για παράδειγμα την αναθεώρηση της οδηγίας Αμφωσόκ και ούτω καθεξής και πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει τρόπος να έχουμε μία σύγκληση απόψεων και να είμαστε υπέρ του σεβασμού των ε, ε, διανοητικών δικαιωμάτων ε, στις ε, ψηφιακές πλατφόρμες. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεισφορά σας. δεν είναι εύκολο να συμπεριλάβουμε όλες τις τροπολογίες σε ένα συμβιβασμό. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε αυτή τη δουλειά που θα οριστικοποιηθεί με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να έχουμε μια συνεκτική γραμμή και να μην ε, έχουμε τεχνητούς ε, και ουτοπικούς ε, συμβιβασμούς. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές και να ακολουθήσουμε τη σωστή άγουσα. Θεωρώ ότι υπάρχει καλή βάση για να τα καταφέρουμε και θα συνεργαστώ με τους Κιώδης. Θα δούμε και τις τροπολογίες που υπέβαλαν όλοι οι συνάδελφοι. Αυτή τη στιγμή, και με αυτό θα ολοκληρώσω κύριο Πρόεδρε, δεν έχω οργανώσει κάποια ημερομηνία για μια συνεδρίαση των σκιωδών νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε εάν δεν υπάρχουν εξαιρετικά φλέγοντα ζητήματα. Ε, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε μια διαβούλευση μεταξύ μας, μεταξύ των ομάδων μας. Δεν χρειάζεται ε, να κάνουμε συνεδρίαση, μάλλον με γραπτή διαδικασία θα καταφέρουμε να συνεννοηθούμε σχετικά γρήγορα. Ε, τουλάχιστον αυτή είναι η απόψή μου. Αν πρέπει όμως και να συνεδριάσουμε επισήμως θα το κάνουμε αλλά νομίζω ότι προς το παρόν μπορούμε να διατηρήσουμε και το προσωρινό χρονοδιάγραμμα, δηλαδή να ψηφίσουμε για τη γνωμοδότηση αυτή στις 3 Μαΐου. Αυτά. Euh, euh, Ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής και τώρα θα ήθελα να ακούσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους συναδέλφους και να απαντήσω και στις ερωτήσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει το λόγο. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη συνάδελφο Λεγκρίπ για τη δουλειά της. Αποτελεί καλή βάση συζήτησης και την ευχαριστώ και γιατί μας είπε ότι είναι διατεθειμένη να ολοκληρώσει αυτή τη δουλειά το συντομότερο δυνατόν για να σεβαστούμε και τις προθεσμίες ε, του χρονοδιαγράμματος ε, και να ψηφίσουμε το Μάιο. Νομίζω ότι υπάρχουν κατάλληλε προποθέσει. Ε, πρέπει απλώς να επεξεργαστούμε λίγο το κείμενο, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν και δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούμε να επακεράσουμε. Να σταθώ σε κάποια πράγματα στα οποία είναι σημαντικά για την πολιτική μου οικογένεια. Τα έχουμε μεταφράσει σε τροπολογίες και η Κωνσταντς μας τις έχει ήδη σχολιάσει. Η πρώτη όσον αφορά τον ορισμό και τις ευθύνες. Ε, είναι δύο θέματα λιλένδετα και είναι σημαντικό πιστεύω ε, για να προστατεύσουμε τους χρήστες και τους καταναλωτές, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και για τους εργαζομένους ε, στον ορισμό της πλατφόρμας. Το αυτό ισχύει και για την ευθύνη η οποία θα πρέπει να ε, προκύπτει από τους κανόνες που θα συντάξουμε. Επίσης, είναι εξίσου σημαντική και η διαφάνεια για τη χρήση των αλγορίθμων. Με τη δυνατότητα, ε, κάτι το οποίο θα δούμε, ε, παρέμβασης και των κρατών μελών για να διορθώσουν τυχόν σφάλματα, εάν υπάρχουν, και για να ε, αποφύγουν και τη διακριτική χρήση των αλγορίθμων. Όπως ε, πολύ σωστά υπενθύμησε η συντάκτρια, είναι πολύ ε, λεπτό το θέμα των προσωπικών δικαιωμάτων και των κεκτημένων αλλά και αυτών των οποίων μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια. Το θέμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ούτως ή άλλως τίθεται σε πολλά από τα θέματα που συζητούμε και σε πολύ διαφορετικά θέματα και σε αυτή την περίπτωση και μάλιστα ίσως σε αυτή την περίπτωση ισχύει περισσότερο από ό,τι σε άλλες. Επομένως θα πρέπει να δώσουμε και τη βαρύτητα που του αρμόζει ε, στο θέμα αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και το θέμα των συνθήκων εργασίας των εργαζομένων. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν ένα διτό αποτέλεσμα. Δημιουργούν νέες ευκαιρίες εργασίας, αλλά καταστρέφουν και πολλές από τις προϋπάρχουσες θέσεις εργασίας. Εμείς λοιπόν δεν θα πρέπει να έχουμε αρνητική στάση, διότι φοβόμαστε αυτή την, ε, φοβούμαστε αυτή τη διαδικασία εξέλιξης της ε, αγοράς-εργασίας, αλλά το πέρασμα από τη μία στην άλλη δραστηριότητα για τους εργαζομένους που σήμερα εργάζονται ή η κατάργηση κάποιων θέσεων εργασίας, η οποία στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από κάποιες άλλες ε, θέσεις εργασίας, χρειάζεται σαφώς καθορισμένους κανόνες. Επομένως, πρέπει για τους εργαζομένους αυτές τις πλατφόρμες ε, το δικαίωμα του ε, συνέρχεσαι και της συλλογικής σύμβασης να επιβεβαιώνεται εκ νόου και να βρίσκεται και πάλι σε αυτή την πορεία των αλλαγών κάποιων εκ των ε, βασικών χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας, ακριβώς για να αποφύγουμε ε, αντιστάσεις οι οποίες θα απορρέουν από την έλλειψη προστασίας ε, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα άλλο ευαίσθητο θέμα, το οποίο έγινε και μείζον θέμα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είναι το θέμα της φορολόγησης πρέπει να υπάρξει ενιαία φορολόγηση και για τις διαδικτυακές και για τις εκτός ε, δικτύου υπηρεσίες. Και αυτό πρέπει να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και πρέπει οι επιχειρήσεις να καταβάλουν φορολογία στη ε, χώρα στην οποία ε, έχουν κέρδη για να αποφύγουμε αρνητικά φαινόμενα όπως αυτά που ε, αποτελούν και το θέμα της ε, έκτακτης επιτροπής για τα Panama Papers ε, ή είχαμε στο παρελθόν άλλες ad hoc επιτροπής για την φορολογία. Διαπιστώσαμε ότι οι αναμαλίες σε θέματα φορολογίας τελικά έγιναν αντικείμενο ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και πρέπει να το αποφύγουμε ευθύ εξ αρχή αυτό το πρόβλημα. Τελευταίο, ένα θέμα εξίσου σημαντικά με τα προηγούμενα, είναι η προστασία των πιο ευάλωτων εργαζομένων, των ατόμων, συγγνώμη, και κυρίω των παιδιών. Ε, ελοχεύουν τεράστιοι κίνδυνοι ε, αν δεν υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου, ε, ρατσισμός, σεξισμός, ε, ε, παρακίνηση της τρομοκρατίας ε, και bullying, εκφοβισμός ε, ανηλίκων. Πρόκειται για θέμα το οποίο φυσικά αφορά και τους ενήλικες, αλλά οι ανήλικοι είναι οι πιο ευάλωτοι και οι πλέον εκτεθειμένοι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα και να προσπαθήσουμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για να τους προστατεύσουμε. Αυτά προς το παρόν. Ε, τώρα, σιγά σιγά όπως θα προχωρούν οι εργασίες ε, που όπω είπα ελπίζω να ολοκληρωθούν και γρήγορα θα ε, δώσουμε και στη συντάκτρια και τη συνεισφορά μας και τις παρατηρήσεις μας για τη συνέχεια τη δουλειά μας. Uh, Thank you very much. Um, σας ευχαριστώ. Αναμένουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, δεδομένου μάλιστα και ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για το θέμα αυτό να μην ξεχνούμε ότι υπάρχει φυστάμενο νομικό πλαίσιο, αλλά ότι η εφαρμογή του δεν έχει γίνει με τρόπο ομοιόμορφο στα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουν προκληθεί έχουν προκληθεί ακριβώ από αυτέ τι διαφορέ στον τρόπο εφαρμογή τη νομοθεσία. Και ίσω θα ήταν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίε για να διευκρινιστεί αυτό. Για παράδειγμα, όσον αφορά το υφιστάμενο καθεστώς για την αστική ευθύνη των ενδιαμέσων που είναι ε, είναι σημαντικό. Πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο ε, τι απαιτείται από μια πλατφόρμα online για να ε, κλείδει τις υποχρεώσεις της εναντί του νόμου. Κάτι άλλο που δεν είναι ξεκάθαρο, μάλλον που θα πρέπει να φροντίσουμε, είναι το ζήτημα της εφαρμογής τη υφιστάμενη νομοθεσία. Για παράδειγμα, για το παράνομο περιεχόμενο υπάρχει ήδη νομοθεσία που υποχρεώνει τι πλατφόρμε αυτή τη στιγμή να αντιληφθούν το περιεχόμενο είναι παράνομο να το κατεβάζουν αμέσω. Ωστόσο, έχουν υπάρξει περιστατικά όπου μια πλατφόρμα χρειάζεται μέχρι και μια εβδομάδα για να ε, κατεβάσει περιεχόμενο αφότου, της, αφότου ενημερώθηκε ότι είναι παράνομο από ένα χρήστη. Επομένως θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ε, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ε, και να ε, φροντίσουμε να εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό και η υποχρέωση notice and take να τα κατεβάζει κανείς στο περιεχόμενο αυτή τη στιγμή ενημερωθεί για τον παράνομο χαρακτήρα του θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει αλληλοεπικάλυψη, δηλαδή να μην υπάρχουν πολλές διαφορετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες να προσπαθούν να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Υπάρχουν άλλες πρωτοβουλίες όπως για παράδειγμα η οδηγία οπτικοκοστικά μέσα ε, ή για το ψηφιακό περιεχόμενο, αλλά δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να τις ε, να, να, να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα με πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες. Αντιθέτω, θα έπρεπε να εστιαστούμε περισσότερο στα νέα προβλήματα, δηλαδή νέες προτάσεις από την πλευρά της Επιτροπής για να αντιμετωπίσει αυτά τα, τα προβλήματα και αυτό θα μπορούσαμε εμείς να το υποστηρίξουμε. Η Επιτροπή, ε, μήπως θέλει το λόγο. Ευχαριστώ από τη Γενική Διεύθυνση Connect και έχω και ε, συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης στα δεξιά μου. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις τροπολογίες, τις οποίες ε, βλέπουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Ε, η προσ... Ε, προσέγγιση της Επιτροπής είναι υπέρ της κοινοτομίας, γιατί αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία που έχουν αυτές οι online πλατφόρμες στην ψηφιακή οικονομία, στην λειτουργία της αγοράς, στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας μόνο στην οικονομία την επιγραμμική, την online, αλλά επίσης και ε, συνήθεις θέσεις απασχόλησης, στην offline αν θέλετε οικονομία, δηλαδή σε μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αξιοποιούν αυτές τις πλατφόρμες ε, για να υποστηρίξουν πλατφόρμες, ε, συγγνώμη, τους πελάτες τους με τρόπους που δεν μπορούσαν πριν και να ανταποκριθούν στην ε, ζήτηση με τρόπους που δεν μπορούσαν πριν. Επομένω, έχουμε μία οικονομία μία η οποία όλο και περισσότερο πηγαίνει προ την κατεύθυνση τη ψηφιοποίηση. Και αυτό είναι ε, καλό και για του καταναλωτέ και για τι επιχειρήσει και για την οικονομία. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, το αναγνωρίζουμε και στην ανακοίνωση, φαίνεται και από τι τροπολογίε, αλλά θα πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία να είναι ουδέτερα από τεχνολογική απόψεω, να αντιμετωπίσουμε μόνο εκείνα τα προβλήματα που όντω υφίστανται, να μην, να μην δημιουργήσουμε ένα υπερβολικό νομικό πλαίσιο ή ρυθμιστικό πλαίσιο, ε, για να μην σταματήσουμε την ανάλυση και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών ε, πλατφορμών. Εμείς θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε την ε, δημιουργία ε, πλατφόρμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, startup, νεοφιών επιχειρήσεων. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε όλα αυτά. Και συχνά έχουμε διαπιστώσει ότι για να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό, δηλαδή το κάθε κράτο μέλο να προσπαθεί να αντιμετωπίζει το και να ρυθμίζει το θέμα διαφορετικά, χρειάζεται να έχουμε μια συνολική προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τώρα συγκεκριμένε τροπολογίε για την ευθύνη, Όπω είπε και η συγγήτρια, ε, προβλήματα, ε, τέτοια θέματα μάλλον αντιμετωπίζονται ήδη σε νομοθετικέ πρωτοβουλίες, άλλε όπως για παράδειγμα η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία. Το ζήτημα του καθεστώτους για την αστική ευθύνη είναι κάτι ξεχωριστό και όντως το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά. Εμείς επιμένουμε στην πρόταση που διατυπώσαμε και στην ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, e-commerce, ε, αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται να προτείνουμε κάποια αλλαγή σε αυτή την οδηγία, αν και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Τον επόμενο μήνα θα δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ενδιάμεση αξιολόγηση της ψηφιακής ε, οικονομίας που έχει διεξαγάγει και κάποια από τα ζητήματα που αναφέρατε θα απαντηθούν εκεί, το Μάιο. Επίσης θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα σε αντικρουόμενα ε, συμφέροντα ή επιδιώξει. Ε, Βεβαίω είναι απαραίτητο το παράνομο περιεχόμενο να κατεβαίνει. Όμω θα πρέπει να ε, διασφαλίσουμε ότι υπάρχει και κάποιο έλεγχο για να μην υποβάλλονται αιτήματα να κατεβαίνει περιεχόμενο το οποίο δεν ήταν παράνομο, ήταν απολύτω νόμιμο. Δεν έχουμε λόγο να δώσουμε τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε επιχείρηση, σε οποιοδήποτε επιχείρηση ε, να λειτουργεί σαν δικαστής και να αποφασίζει από μόνη της ότι ένα περιεχόμενο είναι ε, παράνομο και να απαιτεί το κατέβασμά του. Ε, δηλαδή θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει πάντοτε ένα επίπεδο, μια ισορροπία και μια επιτήρηση, επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων από μια δημόσια αρχή. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντικά και άπτονται του πυρήνα τη πρόταση και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα, όσον αφορά το B2B, έχουν υποβληθεί μια σειρά τροπολογίε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ε, διεξάγει ουσιαστικέ ε, μελέτε. Διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερο μικρές επιχειρήσεις ε, εξαρτώνται από αυτές τις πλατφόρμες. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι υπάρχει έχει ανισότητα στο βάρος που έχει μια μικρή επιχείρηση σε σχέση με τις μεγάλες. Εμείς θα πρέπει να διευκολύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να εστιάσουν στην καρδιά της οικονομικής τους δραστηριότητας. Τα ζητήματα που τίθενται εδώ είναι τα εξή. Τι γίνεται όταν μια μεγάλη επιχείρηση αποφασίζει να κατεβάσει από την πλατφόρμα τη τα προϊόντα μια μικρή χωρί να την ενημερώσει. Ή ο τρόπο με τον οποίο μπορεί να αλλάζουν χωρί προειδοποίηση οι αλγόριθμοι ή τα στοιχεία. Γενικά σε αυτά τα ζητήματα υπάρχει έλλειψη διαφάνεια. Και γενικότερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι ότι δεν έχουν μέσα στη διάθεσή τους δεν, για να αντιμετωπίσουν ε, μια δυσμενή ε, κατάσταση, μια δυσμενή απόφαση. Προσπαθούμε και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρουμε να προετοιμάσουμε το έγγραφο που θα δημοσιοποιηθεί το Μάιο και το οποίο θα απαντήσει σε πολλές από τις ερωτήσεις που θέσατε και στα ζητήματα που αναπτύξαμε εδώ. Σας ευχαριστούμε. Μια ερώτηση για το χρονοδιάγραμμα προς τον εισηγητή, πριν την εισηγήτρια. Έχουμε προβλέψει την ψηφοφορία στην Επιτροπή στην συνάντηση του Μαΐου. Ε, ποια, ποιες ημερομηνίες θα επιθυμιούσατε. Γιατί έχουμε δύο συνεδριάσεις. Μια στην αρχή, αρχές Μαΐου και μια τέλος. 3 και 4 Μαΐου είναι η πρώτη συνεδρίαση και 28-29 Μαΐου η δεύτερη. Η εισηγήτρια Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα και να κάνουμε την ψηφοφορία στην πρώτη. Μάλλον πίστευα ότι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε την ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρία του Μαΐου. Αλλά αν κατάλαβα καλά μου λέτε ότι θα μπορούσαμε είτε στην πρώτη συνεδρία του Μαΐου είτε στη δεύτερη συνεδρία του Μαΐου να κάνουμε την ψηφοφορία. Θα το εξετάσω για να δω τι γίνεται. Να συζητήσω πιθανώς και με τους σκιώδεις, να δω αν προλαβαίνουμε και θα σα ενημερώσω. Okay. Okay, I'm that in order to, to match the IMCO, IMCO timetable. Μα, με, ενημερώνουν από τη γραμματεία ότι εξαιτία του χρονοδιαγράμματο τη Επιτροπή ΙΜΚΟ ε, αναγκαστικά θα πρέπει η ψηφοφορία μα να γίνει στη δεύτερη ε, συνεδρίαση του Μαΐου. συγγνώμη, την πρώτη συνεδρίαση την πρώτη συνεδρία του Μαΐου και διαπιστώνει και η συγκήτρια ότι γι' αυτό προσπαθούσα να προχωρήσω στα γρήγορα έτσι ώστε η ΙΝΚΟ να έχει στα χέρια της το αποτέλεσμα της δικιάς μας εφορίας. Θα ήθελα να απαντήσω και σε κάποια από τα θέματα που έθιξαν οι συνάδελφοι, για τον κύριο Κονφεράτη για παράδειγμα. Θα εξετάσω με προσοχή τις προτάσεις του και το, την τροπολογία που υπέβαλε για την προστασία των ευάλωτων ατόμων και ιδιαίτερα των παιδιών το 76 τροπολογία για τη, τη φορολογία παρά που το γεγονός ότι δεν είναι εμπίπτει ακριβώς στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων το ίδιο και για την τροπολογία 48 που, με την οποία ο κ. Κομφεράτη διατυπώνει τις ανησυχίες που υπάρχουν για τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε αυτές τις πλατφόρμες. Επίσης θεωρώ σημαντικές τις τροπολογίες 66 και 67 για τη διαφάνεια στους αλγόριθμους και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ε, μας διευκρίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κανείς δεν θέλει να αλλάξει το καθεστώς περιορισμένης ευθύνης, δηλαδή το γνωστό ε, άρθρο 14 και 12 έως 15 που ε, δημιουργεί τις οδηγίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο έχει δημιουργήσει το πλαίσιο για την αστική ευθύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και είναι μια συζήτηση την οποία είχαμε και στο πλαίσιο της συζήτησης για την οδηγία για τα πραγματικά δικαιώματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο το γνωρίζουμε. Όμως, μιας και πρόκειται για μια ονομοδότηση ε, την οποία θα υποβάλουμε στην ΙΜΚΟ και την ΙΤΡΕ, θα μπορούσαμε να κάνουμε και κάποιες προτάσεις επί αυτού του καθεστώτος περιορισμένης ευθύνης. Το οποίο έχει θέσμο θετηθεί από τις αρχές του 2000. Ε, αυτά από την πλευρά μου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να συζητάμε αυτό το θέμα. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με το σημείο 14. Ερμηνεία και υλοποίηση της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Το θέμα αυτό έχει δύο συνεισηγητές. Ο ένας είναι ο υποφαινόμενος και ο είναι ο κύριος Κόρμπετ ε, για την ΑΦΚΟ. Να σας ενημερώσω ότι στις 22 Μαρτίου η ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό έκανε την 7η συνεδρίασή της. Η ομάδα έκανε μια ανταλλαγή απόψεων για την απλοποίηση. Ο κύριος ε, Νόρμπερτ Ζάξτετε, εκτελώντα τα καθήκοντα του τμήματιάρχη της ε, Ρέφιτ της Γενικής Γραμματείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η κυρία Κάουφμαν που είναι η συγγήτρια της Επιτροπής μας για την έκθεση ΡΕΦΙΤ ήταν εκεί. Η κυρία Κάουφμαν ε, αναφέρθηκε γενικά στην πρόοδο της Επιτροπής ε, της έκθεσης Ρέφιτ και εστίασε σε οκτώ βασικά θέματα από την έκθεσή της για τα επιτεύγματα ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρακολούθηση ε, των όσων μας είχε προτείνει στις 20 Ιουλίου πέρσι. Αναλυτικά είχαμε την ποιότητα της ε, νομοθεσίας που είναι πολύ πιο σημαντική από την ποσότητα. Η απλοποίηση δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές συνέπειες για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Τρίτον, οι ρήτρες sunset στην νομοθεσία Μπορεί να υπάρχουν, αλλά μόνο με δύο προποθέσει. Ε, μόνο για νομικά πράξεις, νομικές πράξεις οι οποίες είναι περιορισμένες χρονικά και αυτό φυσικά δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της ασφάλειας ε, δικαίου και αν θεωρηθεί απαραίτητο θα ε, επανεξετάζεται η ρήτρα. Επίσης, δεν θα πρέπει να θέτουμε εν κινδύνο το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στα κοινωνικά θέματα, να έχουμε κάποια προγραμματισμένα νομοθετικά ε, σχέδια. Θα πρέπει να υπάρχει σαφή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων από αυτών των θεμάτων. Έκτον, το τεστ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων τους και των εργαζομένων, το, οι εργαζόμενοι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να τη χάνουν τις ίδιες μεταχείρισης και προστασίας με τους εργαζόμενους σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Έβδομο σημείο, το gold plating, ο υπερ, νομικός υπερθεματισμός, να μην υπάρχει επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος. Ε, το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στην υπερβολική νομοθεσία και κανονισμού σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τέλο, όσον αφορά την ανάκληση νομοθεσία, σε περιπτώσει που υπάρχει ανάκληση νομοθεσία ε, ή νομοθετική πρόταση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την άποψή του, η θέση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ζακ Στέτε μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να μειώσει το γραφειοκρατικό, το νομοθετικό μάλλον άχθος μέσω του προγράμματος REFIT και μέσα από αυτό το πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, ελέγχεται συνεχώς προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είναι κατάλληλη για να επιτύχει το σκοπό της και καλύπτει τους βασικούς της στόχους ε, με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Όσον αφορά το, ε, την υπερβολική νομοθεσία και κανονισμούς, ένας τρόπος για να την πατάξουμε είναι να υπάρχει ένας σαφής ορισμός ε, για τις ποιοτικέ και ποσοτικές πληροφορίες. Επεσήμανε ότι αυτές τις μορφές πληροφορίες είναι εξίσου σημαντικές, αλλά τα ποιοτικά στοιχεία είναι μάλλον δύσκολο να βρεθούν από τα κράτη-μέλη. τα από πλευρά Σέμβη η κυρία Βαλεάν ανέφερε ότι θα πρέπει να έχουμε και ποιοτικέ περιβαλλοντικές ε, παρατηρήσεις οι οποίες θα έχουν την ίδια βαρέτητα με τις υπόλοιπες και επίσης ε, ε, τα θέματα της δημόσιας υγείας πολύ δύσκολα μπορούμε να τα ποσοτικοποιήσουμε επομένως καλύτερο θα είχαμε να έχουμε μια προσέγγιση η οποία θα καλύπτει και τις ποιοτικέ πτυχές. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου ενημερωτικά. Δεν ξέρω αν η κυρία Κάουφμαν τώρα θέλει να προσθέσει κάτι. Γνέφει αρνητικά η κυρία Κάουφμαν. Δεν υπάρχει λοιπόν κάτι. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα το σημείο αυτό και συνεχίζουμε με τα κοινά σημεία 15 και 16. που αφορά τους ε, τυφλούς και τις αμφλίωπες και ο λόγος πηγαίνει στον κύριο Άντερσον, ο οποίος είναι η Thank you. This Ευχαριστώ. Έχουμε εδώ δύο ε, προτάσεις που εφαρμόζουν τη σύμφαση του Μαρακές ε, που έχει να κάνει με πρόσβαση σε βιβλία για τυφλούς και άτομα με δυσκολίες στην όραση και με κάποια αναθεώρηση του νόμου περί πνευματικών ε, ε, δικαιωμάτων. Σήμερα, το έχουμε συζητήσει και άλλη φορά το πρόβλημα, είναι ότι όταν έχεις ένα αντίγραφο ενός βιβλίου με μορφή που να είναι προσβάσιμο σε τυφλούς και άτομα με δυσκολία στην όραση, είναι δύσκολο να μεταφέρεις αυτό το αντίτυπο από τη μία χώρα στην άλλη. Έχουμε τα εθνικά σύνορα που δημιουργούν ε, φραγμούς. Είναι κάτι το οποίο κάνει τη ζωή των τυφλών και των ατόμων με τη δυσκολία δύσκολη. Ε, είναι σε ένδια φιλολογική θα λέγαμε. Δεν μπορούν να διαβάσουν βιβλία. Έχουμε 25.000 πιθανούς ε, ωφελούμενους στις ε, φτωχές χώρες που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν βιβλία ε, σε αυτούς τους ανθρώπους. Η, σύμβαση, η συνθήκη της, του Μαρακές ακριβώς αυτό φροντίζει την πρόσβαση σε όλο τον κόσμο των ανθρώπων σε αυτά τα βιβλία. Τώρα υπάρχει μια οδηγία, ένας κανονισμός και είχαμε και την πρώτη συνάντηση της τριμερούς ε, αυτή την Δευτέρα. Έχει γίνει πρόοδος αναφορικά με τους ορισμούς. Η τεχνική ομάδα έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε αυτό το θέμα. Υπάρχει ένα πράγμα όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πω σήμερα. Είναι η νομική βάση. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βρήκε στην τελευταία του γνωμοδότηση σχετικά με τη συνθήκη του Μαρακές ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 207 ως τη νομική βάση για τον κανονισμό. Έτσι πρέπει να βρούμε μια άλλη βάση. Έχουμε λοιπόν να καταλήξει σε μια πρόταση στην τριμερή το άρθρο 114 δηλαδή, που είναι μια καλή λύση θα έλεγα, μπορούμε να δουλέψουμε με αυτή και ελπίζω η Επιτροπή Γιούρη να μπορέσει να συντάξει μια γνωμοδότηση για την αλλαγή της νομικής βάσης το Μάιο, στη δεύτερη συνάντησή μας. Υπάρχουν φυσικά και άλλα θέματα που ε, κρεμούν. Το πιο συγκεκριμένο έχει να κάνει με την αιτιολογική σκέψη 11 της οδηγίας, όπου υπάρχει μια ε, πολύ ηχηρή θέση από την πλευρά του Κοινοβουλίου ότι πρέπει η συνθήκη του Μαρακές να λειτουργήσει και να δώσει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε βιβλία στους ε, τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης με τρόπο δίκαιο και λειτουργικό. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ειδικοί κανόνες και εξαιρέσεις που θα κάνουν τη συνθήκη δύσκολη ή αδύνατη στη χρήση της. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της συνθήκης. Έχουμε λοιπόν ηχηρή θέση εδώ, Ακούγονται ακούγονται ηχηρές απόψεις και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και είμαι αισιόδοξο για το ε, αποτέλεσμα. Μπορώ να συνεχίσω άμα θέλετε, αλλά εντάξει, νομίζω ότι και το ρολόι προχωράει. Η ώρα προχωράει. Δεν θέλουμε να σας αναγκάσουμε να κάνετε κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε αισιόδοξο. Αυτή αυτό το θέμα θέλει η αισιοδοξία γιατί ο χρόνος που έχουμε δαπανίσει δεν αντιστοιχεί πραγματικά στα αποτελέσματα που είναι επίγοντα. For the Κάποια, κάποιο σχόλιο θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο ίσως. Η Κομισιόν δεν θέλει να πάρει το λόγο. Αυτό σημαίνει ότι ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Πάμε τώρα στο σημείο 17, στην ουσία ε, έχει να κάνει με το να ασχοληθούμε και να λάβουμε υπόψη μας συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις για την επικουρικότητα. Τέλος, να σας θυμίζω ότι υπάρχει ε, το απόγευμα ε, στην αίθουσα Γιάν 2Q2 ένα σεμινάριο για την εκπαίδευση των δικαστικών ε, Γιούρι και Λίμπε μαζί και σας ενθαρρύνω να συμμετάσχετε σε αυτό το κοινό εργαστήριο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στη σημερινή μας συνεδρίαση.